οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την Ολομέλεια και θα ε, δημοσιευθούν στα πρακτικά της Ολομέλειας. Έρχομαι τώρα στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ. Παράγραφος 1, σημείο 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τροπολογία 1. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μα. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται σαφώς. Τροπολογία 21 με, προφορι... με ε, ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 των Πρασίνων επίσημο ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης γίνεται δεκτή. Η τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην παράγραφο 13 ή 23 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε έλεγχο εδώ για την τροπολογία 24 και την ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας γίνεται δεκτή 18, τροπολογία 18, υπέρ κατά αποχές δεκτή Εκπίπτει 14 κατά συνέπεια, τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 σε δύο τμήματα και με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Γίνεται δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Πάλι μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι υπέρ κατά αποχές έχει εγκριθεί ερχόμαστε στην έκθεση Μάουρου Θέτω σε ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγχαρητήρια κύριε Μάουρο. Ερχόμαστε στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης <clears throat> με τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Αμερικής, ε, ε, Αφρικής συγγνώμη, σε σχέση με την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε. Ψήφισμα της Γκουε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψήφισμα των Πρασίνων. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το κοινό ψήφισμα τεσσάρων πολιτικών ομάδων. ΕΛΚ, Σοσιαλιστέ, Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι. Ε, τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ενεκρίθη. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 ψήφι υπέρ <clears throat> κατά αποχές γίνεται δεκτή τροπολογία 2 σε 4 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα τέσσερα. υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο για το τέταρτο τμήμα της τροπολογίας 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό το τέταρτο τμήμα. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή με ονομαστική κλίση το σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας γίνεται δεκτό το ψήφισμα Περνάμε στο ψήφισμα στην έκθεση Κασπάρη με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή η έκθεση. Συγχαρητήρια στον κύριο Κασπάρη. Η έκθεση για τον εξυγχρονισμό του, των κρατικών επιδοτήσεων. Ε, χωριστή ψηφοφορία, παράγραφος 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα της 1 σε ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 2 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά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 Παράγραφος 14 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Το σύνολο του ψηφίσματος ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Ερχόμαστε σε ψηφίσματα για τα θύματα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο εφαντουργικών στο Μπαγκλαντές. Ε, τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά από την, ε, το, σκέψη 10. Δύο ταυτόσιμες τροπολογίες. Η 1 και η 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ονομαστική κλίση. <clears throat> Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτό. Μετά την αιτιολογική σκέψη τσε. <clears throat> Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Μόνο η, παρα... Μόνο η τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματο με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. <clears throat> Πέρας. Δεκτό. Ερχόμαστε την, ε, την έκθεση για την μη διάδοση, μη διασπορά των όπλων μαζικής καταστρο, ε, καταστροφής. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτή, γίνεται δεκτό το ψήσιμο και τα άλλα εκτίθουν ως εκ τούτου. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση για την χώρα προέλευσης. Ε, το κοινό ψήφισμα. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό όλα τα άλλα ψηφίσματα εκπίπτουν. Και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Απορρίπτεται, συγγνώμη. Συγγνώμη, λέω πρόεδρος, 11. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Εντάξει, πέρασε. Απορρίπτεται. 12 με ονομαστική κλίση επίσης. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 13 με ονομαστική κλίση. Υπέρ. Ε, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψηφίσατε όλοι, όλες. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το, το συνολικό ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί ψήφι υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Όχι, όχι, όχι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να δω το αποτέλεσμα. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτό. Ευχαριστώ πολύ και καλή όρεξη.